Ευχαριστώ. Δεν βλέπω την κυρία Βρετσιόνοβα. Οπότε κλείνω ε, τις επεξηγήσει ψήφου για αυτό το θέμα και περνάμε στο παράνομο εμπόριο ζώων συντροφίας συντροφιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τελευταία έκθεση για σήμερα. Thank you, Vice President. Ο κύριο Κάλαχερ, πρώτο ομιλητή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για το συγκεκριμένο ψήφισμα και θα ήθελα να ληφθούν άμεσα μέτρα από την Επιτροπή για να αντιμετωπιστεί το θέμα τη παράνομη εμπορία ε, σκύλων και γατών. Ιδιαίτερα το βιομηχανική κλίμακα εκτροφή αυτών των ζώων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα ζώα φυλακίζονται για χρόνια και χρόνια για να παράγουν ε, σκυλα, κουτάβια και γατάκια. Ε, νομίζω πως σαν πολιτισμένη κοινωνία το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να υπάρχει κάποιο είδους ε, καταγραφή για, αυτές, αυτά τις, ε, τα εκτροφία με κάποιο τρόπο να καταγράφονται όλα αυτά ώστε να διέπονται από κάποιους κανονισμούς. Σίγουρα υπάρχει μεγάλο εγκληματικό στοιχείο στην ε, λαθρεμπορία και μετακίν... λαθρομετακίνηση ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έχει επιπτώσεις, αλλά πάνω απ' όλα είναι ένα θέμα βίας κατά των ζώων και ευημερία των ζώων. Και η ίδια η Κομισιόν πρέπει να εξασφαλίσει ότι η εσωτερική μας αγορά διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες και, οι οποίοι να ισχύουν και για αυτές τις, ε, αυτά τα εκτροφία ζώων. κυρία Ντάλη, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, Είμαι πανευτυχής που μπορώ να, και να υποστηρίξω αυτό το ψήφισμα και να καλωσορίσω την πρωτοβουλία που ανελήφθη για αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιά που είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στην Ιρλανδία όπου αρκετοί τα άτομα επιτέλους ε, διώχθηκαν ποινικά επειδή ε, μεταχειρίζονται τα ζώα τόσο φρικτά για δικό τους όφελος και κέρδος. Το θέμα έχει συγκεντρώσει μεγάλη συμπάθεια του ερλανδικού ε, λαού και πραγματικά έχει εντυπωσιάσει γιατί δεν υπάρχουν αρχές, ε, δεν υπήρχαν μάλλον αρχές που να επιβάλλουν ε, την νομοθεσία. Ζητάμε υποχρεωτική ε, καταγραφή και αναγνώριση, ταυτοποίηση των ζώων και επίσης καλούμε την Κομισιόν να απαγορεύσει την εκτροφή και την εμπορία με πρακτικές οι οποίες να είναι εναντίον της ευημερία των ζώων αυτών. Είναι σπουδαίο βήμα μπροστά και γι' αυτό και το υποστήριξα με μεγάλη χαρά. Σα ευχαριστώ πολύ. Επόμενο ο είναι ο κύριος Βέιμερς και έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ. Η μικρή Άστριντ μπήκε στην οικογένειά μας. Είναι ένα υπέροχο σπάνιελ γεμάτο χαρά και ζωή. Ε, Μα είπαν ε, ότι είχε εισαχθεί από τη Σλοβακία και όταν πήγαμε στον κτηνίατρο για μια τακτική ε, εξέταση μα είπε ότι γίνεται συστηματικά απάτη. είτε πρόκειται για τη χώρα προέλευση, είτε για την ημερομηνία γέννησης, έτσι ώστε τα κουταβάκια να μπορούν να, να πουληθούν νωρίτερα από τις 8 εβδομάδες που απαιτούνται ε, για να ελεγχθούν με ασφάλεια αυτά τα ζωάκια και πράγμα το οποίο οδηγεί σε ένα τραύμα για ολόκληρη τη ζωή αυτών των ε, ζώων. Ούτε οι κατάλληλοι εμβολιασμοί είχαν γίνει. Εγώ είμαι υπέρ λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την καταγραφή των ζώων συντροφιά, με την ελπίδα ότι και άλλα ζώα, άλλα σκυλάκια και ζωάκια θα ξεκινήσουν καλύτερα τη ζωή τους από ότι η δική μας Άστριτ. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής ο κ. Πόσπης, Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είμαι ευτυχής που 600 βουλευτές υποστήριξαν αυτό το ψήφισμα <clears throat> κατά του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιά σε ολόκληρη την Ένωση. Πολύ ισχυρό μήνυμα στέλνουμε με την έννοια ότι το Ευρωκοινοβούλιο θέλει να αντιμετωπίσει την λαθρεμπορία αυτών των ζώων και ελπίζω πως η Κομισιόν με βάση το ψήφισμά μας θα ετοιμάσει σαφή μέτρα για να εμποδίσει το να έρχονται, ε, το να εκτρέφονται κουτάβια και γατάκια στην Ανατολική Ευρώπη και να μεταφέρονται σε φρικτές συνθήκες στη Δυτική Ευρώπη για να πουληθούν χρόνο με το χρόνο. Είναι θαρρυντικό ότι το ψήφισμα έλαβε τόσο μεγάλη υποστήριξη και παρακαλώ την Κομισιόν να πάψει να φέρεται, λες και δεν τρέχει τίποτα σε αυτό το τομέα για να αρχίσει να αναζητεί λύσεις. Κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα μόνο του. Είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και ευχαριστώ τους συντάκτες του ψηφίσματος που το υπέβαλαν. Ευχαριστώ. Τώρα έχει το λόγο ο κύριος Στανισλάβ Πόλτσακ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ως ε, συνεισηγητής ε, οπωσδήποτε στήριξα αυτή την πρόταση και χαίρομαι για το ότι μόνο τρεις ε, συνάδελφοι καταψήφισαν. Οπότε προφανώς υπήρχε διακομματική στήριξη. Οπωσδήποτε το θέμα αυτό δεν θα το λύσουν τα κράτη-μέλη μόνα τους. Είναι ένα ζήτημα οργανωμένου εγκλήματος ε, με μεγάλη κερδοφορία. Οι διακινητές ε, δρούν διασυνοριακά. Τα ζώα υποφέρουν, οι καταναλωτές ε, παραπλανούνται, υπάρχει στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς, όλα αυτά. Απογοητεύτηκα κάπως από την δήλωση του Επιτρόπου χτες. Ελπίζω η Κομισιό να συνειδητοποιήσει πόσες χιλιάδες άνθρωποι θέλουν να δράσει η Κομισιόν και ελπίζω η Κομισιόν να το κάνει. Σας ευχαριστώ για την Κουίκιος μπαμπά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το παράνομο εμπόριο αποτελεί μια γάγκρανη την Ευρώπη τα πολλά χρόνια το τρίτο μετά την παράνομη εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Από το 2000 ε, τα κοινωνικά δίκτυα και οι μικρές αγγελίες δείχνουν ότι η κατάσταση επιδεινώνεται. Σύμφωνα με κυβερνητικές οργανώσεις ε, είναι τεράστια η ζήτηση ε, η οποία δημιουργεί κέρδη ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Ε, τα ζώα μεγαλώνουν από τα μεγαλώνουν κλιματικές οργανώσεις σε παράνομες εγκαταστάσεις. Ε, δεκάδες ε, χιλιάδες γατάκια και κουταβάκια αρπάζονται σε πολύ μικρές ηλικίες από τις μητέρες τους, δεν εμβολιάζονται, μεταφέρονται με, σε πολύ κακές συνθήκες αλλού και πολλά από αυτά πεθαίνουν στο δρόμο. Χρειάζεται ένα σύστημα, εναρμονισμένο σύστημα ταυτοποίησης και θα πρέπει να διωχθούν οι πωλήσει. Ε, να απογαρωθούν οι πωλήσει ζών των ζών μέσω ίντερνετ. Σας ευχαριστώ. Και ο τελευταίος ομιλητής, ο κ. Μπότος για το Ρινιό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είχα την ευχαρίστηση πριν από δύο εβδομάδες ε, να οργανώσω μια σχετική συζήτηση στην ε, πόλη μου στη Ρουμανία. Χαίρομαι για το ότι ασχολούμαστε με τους ε, φίλους μας ε, τα κατοικίδια. Πρέπει να σταματήσει το παράνομο αυτό εμπόριο. Πρέπει να σκεφτούμε την ευζοία των ζώων και τη χαρά που φέρνουν στους νέους ιδιοκτήτες. Γίνονται μέλος της οικογένειας. Δεν είναι αντικείμενα που αγοράζουμε. Ε, για τον λόγο αυτό, λόγω του ρόλου που παίζουν στις ζωές μας, νομίζω πως πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα δεν μπορούμε να σταματήσουμε στη ρύθμιση του εμπορίου. Πρέπει να σκεφτούμε τη ζωή των ζώων. Πολλά σκυλιά και γατιά εγκαταλείπονται όταν οι άνθρωποι δεν τα θέλουν άλλο. Είναι η λυπηρή πραγματικότητα και μπορούν να σας δώσουν τις λεπτομέρειες οι σχετικές ΜΚΟ. Πρέπει να το ρυθμίσουμε αυτό. Τι κάνουμε με τα δέσποτα που βρίσκουμε ή νεκρά γατάκια σε σακούλες στο δρόμο. Πρέπει να σκεφτούμε ευρωπαϊκή νομοθεσία για να τα προστατεύσουμε. Τα γατάκια και τα σκυλάκια αξίζουν την ε, προσοχή μας. Πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Μπότος. Τελείωσε η συζήτηση για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. Τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Λούκματς ο οποίος ήθελε να απαντήσει στον τυχερή Μαριανή, με συγχωρείτε, ο οποίος θα ήθελε να απαντήσει σε αυτά που ο κύριος Λούκματς Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είχα προτιμήσει να απαντήσω σε αυτή την προσωπική ερώτηση αμέσως μετά τα όσα είπε ο κ. Γκλουξμαν, αλλά σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο ακόμα και αν είναι τόσο ε, άδειο το ημικύκλιο. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για μία ε, ε, άσχημη ε, παρατήρηση που έκανα. Μίλησα για τη λογική του ε, σφυριού που ορίζει το τέλος του χρόνου αγόρευσης, γιατί αγχώθηκα και δεν μπόρεσα να μιλήσω καθαρά και όπως ε, είχα σκοπό. Δηλαδή, αντί να μιλήσω για εξάλληψη των τροποκρατών, είπα εξάλληψη των επαναστατών. Ε, ζητώ συγγνώμη, πρόκειται όμως για Ισλαμιστές σε αυτή την περιφέρεια και τα τελευταία λέξη τη λέω από την έκθεση του ΟΗΕ που λέει ότι το, το Ιντλίπ είναι το πιο μεγάλο ε, αποθεματικό θύλακας ε, τρομοκρατών σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Ε, έτσι κλείνει η συζήτηση για την ώρα και ε, αναστέλλεται η συνεδρίαση μέχρι τις 3. Καλησπέρα σας συνάδελφοι. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Τα πρακτικά της θεσινής συνεδρίασης είναι στη διάθεσή σας. Υπάρχουν σχόλια. Όχι, οπότε εγκρίνονται. Πρώτο σημείο στην απόψινή ημερήσια διάταξη είναι μια και επίκαιρη συζήτηση. Μια κοινωνική Ευρώπη σε ένα ψηφιακό κόσμο. Θέλω να σα ενημερώσω ότι για αυτή τη συζήτηση δεν θα γίνει catch the και δεν επιτρέπονται μπλε κάρτε. Και ξεκινάμε με τον συντάκτη, τον κύριο Ερτούγκ. Τέσσερα λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ επίτροπε, καταρχάς σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Ε, νομίζω πως οι ψηφιακές τεχνολογίες μας προσφέρουν μια μεγάλη ευκαιρία και δυνατότητες ε, ε, που μπορούμε ε, πολύ εύκολα να τις έχουμε. Παλιότερα ποτέ δεν έχουν μπορέσει τόσο πολλοί άνθρωποι να συμμετέχουν σε μια τέτοια τεχνολογία και να δημιουργήσουν. Δυστυχώς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε όλοι τις απαραίτητες γνώσεις για να αγκαλιάσουμε και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες της ψηφιακής επανάστασης. Εχθές γιορτάσαμε την ημέρα ασφαλέστερου ίντερνετ. Όμως μια μέρα το χρόνο δεν αρκεί Ίσως για να τονίσουμε τη σημασία των ε, δεξιοτήτων στα μέσα ε, ε, αυτά τα τεχνολογικά. Θα πρέπει η εκπαίδευση να εξυγχρονιστεί σε ολόκληρη την Ευρώπη, ώστε να ε, ε, μην υπάρξει χάσμα ψηφιακό στην κοινωνία. Και θέλω να ευχαριστήσω τη Φιλανδική Προεδρία που δίνει, που προσέφερε στους Ευρωπαίους πολίτες ε, δωρεάν πρόσβαση για τα θέματα της, στα θέματα μάλλον της τεχνητής νοημοσύνης. Μπορεί αυτό να έχει τεράστιο όφελος για το κόσμο και για τις κοινωνίες. Πρέπει όμως εμείς να το σκεφτούμε καλύτερα γιατί οι πολιτικές απασχόλησης και οι κοινωνικές πολιτικές θα πρέπει να συμβαδίσουν με την ψηφιοποίηση των αγορών εργασίας. Χρειάζεται ένα κοινωνικό σύμφωνο για τον νέο αυτό κόσμο που θα περιλαμβάνει κατώτερους μισθούς, θα ενισχύει τις συλλογικέ διαπραγματεύσεις και ιδιαίτερα και το δικαίωμα αποσύνδεσης. Ε, Επίση, χρειάζεται να δημιουργηθούν δίκαιε συνθήκε εργασία ε, για του εργαζόμενου, είτε είναι επιγραμμικά είτε όχι και πρέπει να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους ε, γίγαντες της ε, πληροφορικής που καταχρώνται την αγορά. Επίσης θα πρέπει να καταβάλλονται οι φόροι εκεί όπου ε, δημιουργούνται τα κέρδη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να φτιάξει ένα νέο πλαίσιο για τη τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ συμπεριλαμβανομένων των, εγγυήσεων για την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το λευκό βιβλίο στην επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να χειριστεί αυτό το θέμα όσον αφορά την ασφάλεια και την ευθύνη. Και οι αλγόριθμοι δεν θα πρέπει να διέπονται από προκαταλήψεις, θα πρέπει να κάνουν διακρίσεις επί τη βάση φύλου ή εθνότητας και λέμε όχι τεχνητή νοημοσύνη χωρίς ε, διοντολογία.